Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ώρα να ξεκινήσουμε, γιατί πρέπει να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και όπως ε, ξέρετε δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα και θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο Ανδρουκάητη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η Κομισιόν έχει εγκρίνει χθε τα κριτήρια για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες για να εξασφαλίσει λοιπόν ότι υπάρχει μια κατάταξη για τα προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτήρα ενδοκρινικών διατρακτών. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και για την ανθρώπινη και την ζωική υγεία, αλλά και για την υγεία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα την διαθεσιμότητα του κυρίου Επιτρόπου να μας παρουσιάσει τα προτινόμενα κριτήρια στη σημερινή μας συνεδρίαση και προσβλέπω στο να ακούσω και τις λεπτομέρειες της πρότασης αυτής και τα επόμενα βήματα της, Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ και σας δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα ψήφισμα που ζητά από την Κομισιόν να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, με το να παρουσιάσει επιστημονικά κριτήρια για την ε, διακρύβωση του αν ένα προϊόν είναι ενδοκρινικός ε, διαταράκτη. Έχω λοιπόν αυτή τη ε, μεγάλη χαρά να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου να παρουσιάσω τις θέσεις της Κομισιόν ενώπιον του Κοινοβουλίου. Παρουσίασε λοιπόν η Επιτροπή τα επιστημονικά αυτά κριτήρια στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και των ε, νομοθετημάτων για τα βιοκτώνα. Σας λέω και πάλι. Στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των ε, εδαφών και για τα βιοκτώνα προϊόντα. Τα επιστημονικά αυτά βασίζονται στους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Λέει αυτός ο ορισμός. Μια χημική ουσία είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, αν πρώτον έχει αρνητικά αποτελέσματα και δεύτερον, αν αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται από ενδοκρινική λειτουργία. Επομένως, η ανακοίνωση της Κομισιόν δεν περιλαμβάνει μονάχα αυτά τα επιστημονικά κριτήρια, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διακρύβωση του αν κάτι είναι ενδοκρινικός διαταράκτη. Είναι απαραίτητο αυτή η διαδικασία διακρύβωσης να χρησιμοποιεί επιστημονικά κριτήρια, να χρησιμοποιεί μια <clears throat> αντιμετώπιση η οποία σταθμίζει τα, τις ενδείξεις και τα στοιχεία στη διαδικασία μας και εφαρμόζει αυτή την συστηματική αντιμετώπιση. Εμείς έχουμε πάρει μια μετριοπαθή ε, προσέγγιση θέλοντας να έχουμε ένα ε, εύλογο σταθμισμένο επίπεδο στοιχείων και όχι οριστικά στοιχεία. Δηλαδή σε περίπτωση ε, αμφιβολίας θα δρούμε βάση της αρχής της πρόληψης με μια προληπτική προσέγγιση. Η Κομισιόν επίσης ενέκρινε μια ανακοίνωση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που παρουσιάζει το πλαίσιο το ρυθμιστικό. Όπως ξέρετε υπάρχουν πολλά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που αφορούν τους ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες. Το RIS, τα οδηγίες για την ποιότητα των υδάτων, για τα καλλιντικά κτλ. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει και μια πλήρη έκθεση αντικτύπου. Η απόφαση της Κομισιόν λοιπόν να οριστικοποιήσει αυτήν την ε, έκθεση αντικτύπου έτυχε επικρίσεων και από μέλη της Επιτροπής σας. Αλλά πιστεύω ότι ήταν σημαντικό το έργο αυτό για να δώσει τη δυνατότητα στο Σώμα των Επιτρόπων να πάρει μια καλώς πεπληροφορημένη απάντηση και απόφαση για το σημαντικό αυτό ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο και τα κάτι μέλη θα είναι επίσης σε θέση να επωφεληθούν από αυτό το έργο. Προκαταλαμβάνω το ερώτημα το οποίο θα μπορούσατε να μου πείτε, να μου δώσετε, Θέλω να πω ότι η απόφαση της Κομισιόν βασιζόταν σε επιστημονικά δεδομένα και όχι κοινωνικο-οικονομικές ε, θεωρήσεις. Έχουν δημοσιευτεί όλα αυτά τα στοιχεία στην ε, ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ε, Κομισιόν για να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη διαφάνεια. Έχουμε το πιο προστατευτικό και αυστηρό πλαίσιο για την προστασία που βασίζεται σε στεναρά επιστημονικά δεδομένα. Αυτό οφείλεται και στην πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έγκριση μια ουσία προποθέτει ότι έχει γίνει μια πλήρη αξιολόγηση από εμπειρογνώμονε των κρατών μελών και έλεγχο ομοτήμων από την ΕΦΣΑ ώστε να ανταποκρίνονται στον κατάλογο των ε, χρήσεών τους και εφόσον εξασφαλίζεται ότι δεν έχουν αντικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη τη ζωική υγεία ή το περιβάλλον οι κανόνες για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες έχουν εισαχθεί πριν από λίγα χρόνια με ενδιάμεσα κριτήρια σε μια εποχή που δεν ήταν δυνατόν να καθορίσουμε επιστημονικά τα κριτήρια αυτά για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών. Η συζήτηση για τα θέματα αυτά έχει συζητήσει τα τελευταία χρόνια μεταξύ επιστημόνων και πολιτικών. Προσωπικά Έχω συναντήσει και έχω ακούσει τις απόψεις πολλών επιστημόνων από πολύ διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, <clears throat> γιατί κάθε άποψη έχει μια διαφορετική φρασιολογία και λογική και μας βοηθάει να καταλάβουμε τη μεγάλη πολυπλοκότητα του αντικειμένου. Νομίζω ότι είναι και χάρη στις κοινέ προσπάθειές μας που έχουμε ξεκινήσει αυτές τις συζητήσεις, ώστε έχει για πρώτη φορά διατυπωθεί μια επιστημονική συνένεση 23 διεθνούς φήμης ε, επιστημόνων τον Απρίλιο του 2016. Έχουμε λάβει υπόψη αυτή τη γενική συνένεση ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε τα κριτήρια που έχουμε παρουσιάσει. Επιπλέον, εμείς προτείνουμε να υπάρξει και μια εξαίρεση για την προστασία για, φυτο, για προστασία φυτικών προϊόντων ώστε να αντανακλά τις επιστημονικές γνώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε όλες τις επιστημονικές πληροφορίες για την έκθεση και τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Η Κομισιόν θα πρέπει να μια, πάρει μια απόφαση για αυτή την εξαίρεση επί τη βάση όλων των στοιχείων. Η έκθεση μονάχα σε αυτά τα προϊόντα δεν είναι αρκετή για να δοθεί σαφήνεια στο επίπεδο κινδύνου σε σχέση με αυτήν την ουσία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλες ε, εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν για τα κριτήρια σε σχέση με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Εκπροσωπούν αυτές οι εναλλακτικές απόψεις θέσεις κατών μελών ή εμπλεκομένων ή και ε, επιστημόνων. Ορισμένοι λένε ότι θα πρέπει να προσθεθεί η ενεργητικότητα των ουσιών αυτών και να υπάρξει και αυτό στον ορισμό του ΠΟΕ, πέραν του ορισμού της ΠΟΕ. Άλλοι θέλουν να έχουν κριτήρια που να βασίζονται σε διαφορετικέ κατηγορίες επί τη βάση του επίπεδου των στοιχείων και των ενδείξεων που υπάρχουν. Η Κομισιόν δεν έκανε τίποτα από αυτά <clears throat> για τον εξή λόγο. Πρώτα απ' όλα, η επιστημονική συνένεση που ανέφερα προηγουμένως καταδεικνύει ότι το επίπεδο ενεργητικότητος μιας ουσίας δεν πρέπει να είναι τμήμα της, ε, του ορισμού ενός ενδοκρινικού διαταράκτη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αξιολογούμε το κίνδυνο που μπορούν να προκαλέσουν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Βασιζόμαστε λοιπόν στις επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες και δεν χρησιμοποίησαμε την ενεργητικότητα μιας ουσίας, τον χαρακτήρα της ως ενεργό. Για την κατηγοριοποίηση επίσης η Κομισιόν δεν θεώρησε ότι το να έχουμε διαφορετικές κατηγορίες σε σχέση με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, σε σχέση με την ενδεχόμενη ιδιότητά τους ως ε, διαταρακτών, με αυτόν τον τρόπο δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη να καθορίσει τι θα πει πραγματικός ενδοκρινικός διαταράκτης, όχι ένας δυνητικά ή ίσως διαταράκτης. Η χρήση των κατηγοριών στην οδηγία για τα βιοκτώνα και τα ε, παραστοκτώνα θα μείωνε την ασφάλεια δικαίου. Η νομοθεσία λοιπόν, και θέλω να το τονίσω, τη νομοθεσία αυτή που ψήφισε το Κοινοβούλιο δεν δίδει εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε πιθανά ή πολύ πιθανά ή πολύ, πολύ πιθανές μάλλον ή υποψιαζόμενες περιπτώσεις ενδοκρινικών διαταραχτών. Δε έτσι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε σύγκριση χωρίς να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Σε σχέση με τη δυνατότητα να κρατήσουμε τα προσωρινά κριτήρια τα οποία αυτή τη στιγμή ισχύουν στην νομοθεσία για τα βιοκτώνα και τα παραστοκτώνα, αυτό απερίφθη γιατί αυτά τα, κριτήρια δεν είναι κατάλληλα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί βουλευτέ, τα χθεσινά κριτήρια βασίζονται στου ορισμού του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεία. Είναι κατάλληλα, είναι επιστημονικά και δίνουν εγγύηση του υψηλότερου επίπεδου προστασία τη ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλοντο. Για την προστασία των εδαφών και την αντιμετώπιση των βιοκτώνων ουσιών. Τα κριτήρια τώρα αυτά βέβαια θα πρέπει να εγκριθούν με την απαραίτητη διαδικασία. Θα πρέπει να συζητηθεί η κατεξουδότηση πράξη για τα βιοκτώνα από εμπειρογνώμονε των κρατών μερών και μετά θα εγκριθεί από την Κομισιόν. Η ρύθμιση για τα παραστοκτώνα θα ε, εξεταστεί και θα ψηφιστεί στη μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και οι δύο αυτέ αποφάσεις θα υπόκεινται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι συνεργασίε λοιπόν θα είναι κέρια και ελπίζω ότι θα μπορέσω να βασιστώ στην υποστήριξή σα για την έγκριση των κριτηρίων αυτών που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό ρόλο για την προστασία τη υγεία και του περιβάλλοντο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν επίση και για την χημική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα αντιμετωπιστούν και να εξεταστούν και από άλλε χώρε. Με τον τρόπο αυτό το εθνιστικό σύστημα για αυτές τις ουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι το πρώτο σύστημα το οποίο θα σπίσει κριτήρια για την ε, αναγνώριση των ενδοκρινικών διαταρακτών και έτσι θα γίνουμε πρωτοπόροι σε αυτό το σημαντικό τομέα. Η ΕΦΣΑ και η Υπηρεσία για τα Χημικά, η ΕΚΑ, έχουν ήδη ξεκινήσει να κοιτούν ορισμένες συγκεκριμένες ουσίες για να μπορέσουν να προετοιμάσουν την εφαρμογή των νέων κριτήριων από τη στιγμή που θα εγκριθούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ξέρω ότι θα έχετε ερωτήματα. Θέλω να σταθώ σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε και χθε από τον Πάβελ Πότς. Ο Πάβελ Πότς μας ρώτησε γιατί προτείνουμε κριτήρια μονάχα που αφορούν την ανθρώπινη υγεία. Αυτό σημαίνει ότι πολύ λίγες ουσίες θα κατονομαστούν ως ενδοκρινικοί ε, διαταράκτες. Και είπα ότι αυτό δεν συνάδει με τον ορισμό του ΠΟΕ. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι μια παρεξήγηση και θέλω να τη διευκρινίσω. Προτείνουμε κριτήρια για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και για το περιβάλλον. Στην ε, κατεξοδότηση πράξη για τα βιοκτώνα έχετε τον τομέα Α που είναι η ανθρώπινη υγεία και τον τομέα Β για όργανα τα οποία δεν είναι αντικείμενο στόχευση. Έχουμε επίση και τα μέτρα για προϊόντα προστασίας φυσών. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι για να εφαρμόσουμε αυτά τα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλε τι απαραίτητε εμπειρογνωμοσύνε που καλυπτούν και του δύο τομείς. Όταν λέμε λοιπόν για τα ε, παραστοκτόνα και τα βιοκτόνα, ξέρουμε ότι μιλάμε για το περιβάλλον. Προφανώς αλλά το περιβάλλον αυτό επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία και φυσικά και τη ζωική υγεία, την υγεία των ζώων. Επίσης ένα θέμα ήταν ότι τα κριτήρια βλέπουν μονάχα, λαμβάνουν υπόψη μόνο τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι πολύ λίγες ουσίες θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ως ενδοκρινικοί ε, διαταράκτες. Και το ερώτημα αυτό ήταν λοιπόν μήπως χρησιμοποιείται τον πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ειδικά χειρίδια αυτό είναι μια παρεξήγηση. Δεν βλέπουμε μόνο τα γνωστά αποτελέσματα, λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα και θα αξιολογούμε με μια προσέγγιση σταθμισμένης, σταθμισμένων ενδείξεων. Και δεν μιλάω μονάχα για αποδεδειγμένα προϊόντα, που είναι διαταράκτες. Χρησιμοποιούμε όλες τις ε, ε, μελέτες, τις μελέτες in vitro, τις μελέτες σε ζώα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τους ε, διαταράκτες. Γενικά την επιστημονική λογοτεχνία. Προσπαθούμε λοιπόν προσπαθούμε να δούμε και τη βιολογική ε, πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της ε, αρχής της πρόληψης. Όταν υπάρχουν νέα στοιχεία θα τα συμπεριλάβουμε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο. Καταρχάς, οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων θα λάβουν το λόγο, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί δεν έχουμε σήμερα πολύ χρόνο. Η Φρασάς Γκροστέτ θα ξεκινήσει από πλευρά του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε και μας ε, δώσετε αυτές τις πληροφορίες. Ε, θέλω να σας πω ότι με καθησυχάσατε εν μέρη. Ε, παραμένω ανήσυχη. Καθησυχάστηκα γιατί άκουσα αυτά τα κριτήρια. Ουσιαστικά είναι η ίδια με αυτά που προβλέπει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και αυτό είναι, συνενετι... είναι κάτι που βρίσκει σύμφωνη την περισσότερη ε, την πλειοψηφία της ιατρικής κοινότητας. Όμως όταν μιλάμε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες πρέπει να δούμε τον ορισμό με πολύ προσοχή γιατί έχουμε ένα σύστημα παρεκκλήσεων με βάση την έκθεση και τους κινδύνους. Αν κατάλαβα καλά διαβάζοντας το έγγραφό σας, ε, μια ουσία μπορεί να αναγνωριστεί ως ενδοκρινικός διαταράκτης, αλλά να την χάνει παρέκκληση στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτώνα, επειδή ο κίνδυνος ποτέ ότι θα είναι αμεληταίος. Αυτή η αρχή της παρέκκλησης όμως δεν λαμβάνει υπόψη τα λεγόμενα αποτελέσματα κοκτέιλ. Δηλαδή βασιζόμαστε στην αξιολόγηση ε, του κινδύνου αλλά τελικά ε, Αντί για danger μιλάμε για risk. Βασίζεται η αξιολόγηση στο κίνδυνο danger, όπως προβλέπει ο κανονισμός για Με, το, με αυτές όμως τις εξαιρέσεις βάσει ανάλυσης του risk, εκεί έχουμε πρόβλημα. Και από τη σελίδα 5 λέτε ότι δεν θα δημιουργηθεί σύστημα κατηγοριών, που εγώ όμως θεωρώ ότι είναι χρήσιμο. Στη σελίδα 6 μας λέτε ότι είναι δύσκολο να ορίσουμε κατόφλια ε, έκθεση, ασφαλούς έκθεση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε παρεκκλήσει με βάση έναν αμεληταίο, ένα αμεληταίο ρίσκο ε, και στην ίδια σελίδα το κριτήριο της ισχύω ε, το, δεν το λαμβάνετε υπόψη. Αλλά λέτε ότι για την αξιολόγηση του ρίσκου μπορούμε να το μελετήσουμε αυτό το κριτήριο. Θα μπορέσουμε, πιστεύω, να καταλήξουμε σε συμβιασμό, αλλά νομίζω ότι έχετε κάνει το μισό δρόμο. Δεν λαμβάνετε πραγματικά μια απόφαση και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα συνονθήλευμα από διατάξει ε, και αυτό ε, σίγουρα που πρέπει να έχουμε υπόψη μα είναι η υγεία των καταναλωτών. Κύριε Δημοσιακή, ευχαριστώ. Thank you, Chair, and, uh, από τους Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ήρθατε εδώ και μας ε, ενημέρωσε για αυτά τα κριτήρια. Το είχατε υποσχεθεί να το κάνετε πριν από τις θερινές διακοπές. Ευχαριστώ για τις ε, απαντήσεις που μου έχετε δώσει, μας έχετε δώσει. Όμως, προτείνετε αυτά τα προσωνά κριτήρια. Και λέτε ότι ετοιμάστε για άλλα νομοθετήματα άλλα ενδιάμεσα κριτήρια. Αλλά γιατί δεν έχετε εφαρμόσει οριζόντια κριτήρια για να αντιμετωπίσετε την πολυπλοκότητα του προβλήματο, καλλιτικά, χημικέ ουσίε κτλ. Με εξέπληξε ιδίω μια δήλωση στην σύνοψη στη σελίδα 7. Για τον καθορισμό. Δυστυχώ δεν μιλάει στο μικρόφωνο, μιλήσει και δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Uh, uh, Έχω διαβάσει έγγραφα του Κοινοβουλίου Δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφεται ακριβώς εδώ σε αυτό το έγγραφο. I want mention today... Μιλήσατε για μικρέ αλλαγές στη διατύπωση. Αλλά δεν είναι μικρές, για μένα είναι ουσιαστικέ. Στο παράδειγμα 2. May cause adverse effects, λέει no to have adverse effects. Και μιλάτε για τις ιδιότητες ε, ενδοκρινικού διακράκτη πάλι με μια διαφορά στη διατύπωση. Επίσης, μιλάτε για αμεληταία έκθεση και μετά για αμεληταίο ρίσκο. Από hazard-based πάμε σε risk-based. Αλλά εγώ νόμιζα ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η προσέγγιση για να μιλάμε για κίνδυνο, hazard. Πώς αιτιολογείται την αλλαγή αυτή σε σχέση με αυτά που ενέκριναν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και πόσο ε, συνάδει αυτό με την απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, μπορεί να αλλάξει και τα λοιπά και τα λοιπά με βάση το άρθρο 290. 90. Άρα δεν ξέρω, ευθυγραμμίζεται λοιπόν αυτό με αυτά που λέει η απόφαση ε, που σας ε, ανέφερα. Και αν ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αν έχετε επιλέξει τέλο πάντων για κάποιο λόγο. Αυτή την αλλαγή hazard-based σε risk-based, πώς αυτό θα συνεισφέρει στην προστασία της υγείας των Ευρωπαϊκών πολιτών και στην προστασία των καταναλωτών. Υπάρχουν καρκινογόνα, γενοτοξικά και παραμένουν κατηγορίες και η προσέγγιση εξακολουθεί να βασίζεται στον κίνδυνο χάζαρτ και όχι στο ρίσκο. Ενώ εδώ αλλάζουμε στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Uh, η Τζούλη Γκέρλινγκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Κύριε Επίτροπε, φαντάζομαι ότι κάποιους ε, τους χαροποιείτε σε κάποια σημεία. Ε, όλοι μας με κάποια συμφωνούμε, με άλλα όχι. Θα σας δώσω τη δική μου προσωπική εντύπωση. Χαιρετίζω τον ορισμό που ε, είναι ευθυγραμμισμένος με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για να έχουμε συνέπεια με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης θετικό είναι που εστιάζεται στην σχέση, στην αιτιώδη συνάφεια ε, της δράσης και της ανεπιθύμητης ενέργειας. Πολύ σημαντικό να γίνεται η διάκριση η πραγματική ενδοκρινική διατάξη πρέπει να διαχωρίζεται από άλλες ουσίες που απλά επιδεικνύουν μια δράση ενδοκρινικής διαταραχής. Καλό είναι επίσης ότι για ύποψη ενδοκρινικούς διαταράκτες δεν εισάγεται κατηγορία. Είναι καλό αυτό. Επίσης, σε σχέση με τι επιθυμητέ ενέργειε που είναι έμεσε συνέπειε άλλων τοξικών αποτελεσμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη για την αναγνώριση αντοκρινικών διδακτών. Άρα εστιάζουμε στο ειδικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επίση, καλό είναι που εστιάζεται σε επιστημονικέ αποδείξει. Έτσι τα κριτήρια θα εφαρμόζονται με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο και θα έχουμε ψηλό επίπεδο προστασίας. Αυτά είναι τα θετικά. Υπάρχουν και αρνητικά. Με απογοητεύει το ότι τα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στο λεγόμενο biological plausibility και όχι σε ε, τεκμήρια διάστα. Λέτε ότι είναι δύσκολο. Δύσκολη είναι γενικά ε, το πώς μπορούμε να τα αποδείξουμε όλα αυτά. Αλλά δεν θα πρέπει τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε. Θα το συζητήσουμε για καιρό αυτό το biological plausibility. Σίγουρα υπάρχουν κενά γνώσεων. Ελπίζουμε να γεμίζουν σιγά σιγά αυτά τα κενά. Οπότε ελπίζω να μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για την ισχύ, το πότενση, δεν θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στον ορισμό ενός ενδοκρινικού διατάκτη, αλλά μόνο στην αξιολόγηση του κινδύνου. Τώρα έχουμε όμως το κριτήριο. Και υποτίθεται ότι το αναθετικό πλαίσιο είναι πλήρες. Μόνο σε παρεκκλήσεις μπορούμε λοιπόν να το βάλουμε αυτό το κριτήριο. Είμαι ίσως ε, αντίθετα από αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ. Εγώ θέλω να μπει στην νομοθεσία οι παρεκκλήσει. Είναι εξαιρέσει εκφύσεως. Αντί να εφαρμόζουμε συστηματικά λοιπόν τις εξαιρέσεις που θα είναι και πολλές και να μην έχουμε τελικά ένα ε, μοσαϊκό και ένα πολύ κακό κανονισμό τελικά λόγω των εξαιρέσεων και όλων αυτών των αξιολογήσεων κινδύνων, καλό θα ήταν να έχουμε μια βάση, έναν βασικό κανονισμό. Thank you very much. Miss... ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, την προηγουμένη εβδομάδα, λέει κύριε Χάζεκάμπ, το Κοινοβούλιο έδωσε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το καθήκον της όσον αφορά τους ε, διαταράκτες. Το 2013 εσείς αναλάβατε την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων αλλά και του περιβάλλοντος. Προστασία από αυτά τα φάρμακα. Και πέρασαν τρία χρόνια και έρχεστε και μας μιλάτε για το κριτήριο του κινδύνου. Έχουμε εκατοντάδες μελέτες, ομοτήμων κλπ. Οπότε ακόμα ε, κατέληξαν αυτές οι μελέτες και οι χαμηλότερες δόσεις αυτών των φαρμάκων και ουσιών έχουν σοβαρές συνέπειες για έμβρια και για τους ανθρώπους γενικότερα. Τι γίνεται με τα οικονομικά κριτήρια, τι γίνεται με ε, τον, τη στρέβλωση του ορισμού του Οργανισμού Υγείας. Τι γίνεται με την αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Έτσι δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία. Και έχουμε και όλα αυτά τα πειράματα με τα ζώα. Μα δεν χρειάζονται γιατί αφού είπαμε ότι όλες οι μελέτες κατέληγουν ότι ακόμα και οι χαμηλές δόσεις έχουν βλαβερά αποτελέσματα. Παίζετε μαζί μας. Παίζετε παιχνιδάκια με την υπόθεση υγεία. Το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να εγκρίνει μια τέτοια πρόταση. Θα πρέπει να μην είμαστε συνένοχοι σε αυτό που γίνεται. Ήδη έχει αποφανθεί ε, κατά των προτασιών σας στο δικαστήριο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει το καθήκον του. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Επίτροπο, λέει ο κύριος Σέκχαλ. Μίλησατε για τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν. Εγώ ξέρετε χθε παρακολούθησα την συνέντευξη τύπου και υπήρξαν πολλέ ερωτήσει από πλευράς δημοσιογράφων σε σχέση με τα πειράματα που γίνονται σε ζώα και είπατε δεν θα απαντήσω επ' αυτού, το είπατε τρεις φορές, μήπως θα έπρεπε να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι πολιτικά θέματα που μπορείτε να τα προσπεράσετε, είναι θέματα τεχνικά. Κάνουν το καθήκον στη δημοσιογραφία που τα ρωτάνε. Πάντως εδώ πέρα έχουμε δύο αντιρρήσεις. Πρώτα-πρώτα ε, είναι θέμα περιεχομένου και επίση το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την νομοθεσία. Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο, αυτό το οποίο κάνετε είναι το εξής. Για να αποδείξετε τι κάνει διαταράκτης λέτε ότι θα πρέπει να έχει ε, εγνωσμένα αποτελέσματα ε, για τα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό ε, αποτελεί μια στρέβλωση του, θα, τι θα πει αρνητικό αποτέλεσμα λέμε κατά πόσο είναι γνωστό κάτι ή όχι, αλλά έχουμε και την κατηγορία Β, όπου εκεί λέμε ότι επί τη βάση των πειραμάτων σε ζώα υπάρχουν, υπάρχει πιθανότητα αρνητικών αποτελεσμάτων. Άρα είναι θέμα απόδειξης. Όμως αυτό το οποίο κάνετε είναι περιορίζεται λοιπόν τον κύκλο των διαπιστώσεων. Ε, λέτε ότι σέβεστε τους επιστήμονες, να σας πω τι λένε οι επιστήμονες. Και η, εταιρεία των ενδοκρινολόγων που είναι πιο μεγάλος ε, φορέας επ' αυτού κατέληξαν στο ότι τα κριτήρια της Επιτροπής είναι υπερβολικά στενά και δεν προστατεύουν τον κόσμο από αυτές τις ουσίες από αυτά τα φάρμακα. Ε, αφού αυτό λέει ναι, οι επιστήμονες ε, τότε έχετε πρόβλημα με αυτές τις προτάσεις. Λέτε όχι αλλά θα πρέπει όμως να απαντήσετε Κάνουν λάθος αυτοί οι επιστήμονες. Γιατί ε, στενεύεται τόσο πολύ τον ορισμό και τα κριτήρια. Επίσης, επί της διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει μόνο κάποια νομοθεσία που ήδη ισχύει εάν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση περί τούτου. Εσείς εδώ αλλάζετε το παράρτημα και λέτε εκτός εάν υπάρχει έκθεση και το κάνετε εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους. Από το exposure το, κάνετε risk. Έκθεση και κίνδυνος. Αυτό είναι απόφαση πολιτική. Δεν έχει καμία σχέση με αλλαγή επιστημονική, τεχνοκρατική. Είναι πολιτική κίνηση αυτή και δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο και για να ισχύσει κάτι τέτοιο χρειάζεται συνομοθεσία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αυτό που κάνατε δεν επιτρέπει το κάνει η Επιτροπή. Επομένω, εμεί για λόγου περιεχομένου αλλά και τύπου δεν θα δώσουμε το πράσινο φω στι προτάσει. Ευχαριστώ κύριε Αντωνάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Σε μια ανακοίνωση, ο πρόεδρος Γιούνκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρώτο σύστημα στον κόσμο που καθορίζει επιστημονικά κριτήρια για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες με νομοθετική πράξη. Αυτό όμως ξεχνά λιγάκι ότι ο κανονισμός αυτός ακολούθησε την καταδίκη της Κομισιόν τον Δεκέμβριο 2015 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν είχε καθορίσει έγκαιρα αυτά τα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια βασίζονται σε αυτά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είναι μια αξιόπιστη βάση. Βέβαια δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη την έννοια της ενεργητικότητος που θα πρέπει να περιλαμβάνει και κατόφλια. Επίσης, η εξαίρεση προβλέπει μια προσέγγιση με ανάλυση κινδύνου, δηλαδή της έκθεσης του πληθυσμού. Θα πρέπει να γίνει και μια αξιολόγηση κινδύνου πριν από οποιοδήποτε κανονισμό για μια ουσία. Επομένως, δεν έχουμε σταματήσει να περιμένουμε να έχουμε χρόνο αναμονής για να υπάρξει προστασία εναντί αυτών των ουσιών. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είχε παρουσιάσει τον ορισμό του πριν από 14 χρόνια. Οπότε η ανάγκη να υπάρξει μια μελέτη αντικτύπου <clears throat> δεν είχε σαν στόχο παρά μόνο να καθυστερήσει τη ρύθμιση και να βοηθήσει τα λόμπι, δυστυχώ. Τέλο, η Κομισιόν έδωσε εντολή στην ΕΦΣΑ και την ΕΚΑ να αξιολογήσουν ορισμένε ουσίε οι οποίε μπορούν να είναι ενδοκρινικοί διαταράκτε. Επί τη βάση των χθεσινών κριτηρίων. Μα θυμηθείτε ότι η ΕΦΣΑ θεώρησε ότι η γλυφοσάτη είναι κατά πάσα πιθανότητα μη καρκινογόνο σε αντίφαση με την άποψη του ΣΥΡΚ, του οργανισμού που εξαρτάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχω δύο ερωτήματα λοιπόν να σας δέσω κύριε Επίτροπε. Την επόμενη φορά που θα υπάρξει μια διαφωνία απόψεων μεταξύ της ΕΦΣΑ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ποιον θα πιστέψετε. Και δεύτερο ερώτημα, αν η αρχή της πρόληψης επικρατεί και υπερέχει όπως είπατε, μήπως τα κράτη-μέλη τα οποία είναι πιο επιφυλακτικά και θέλουν να απαγορεύσουν ορισμένε ουσίες μπορούν να το κάνουν χωρίς προβλήματα και χωρίς κίνδυνο να ε, θεωρηθεί ότι θέτουν προσκόμματα στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος, Κύριε Σπαρνιώ. Κύριε Επίτροπε, θέλω να χαιρετήσω την παρουσία σας και την παρουσίαση που κάνετε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό είναι πολύ καλό, είναι μια καλή ε, πρόθεση από τη δική σα πλευρά και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό 24 ώρε μετά μια ανακοίνωση τη Κομισιόν να υπάρχει συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά θέλω να τα υπογραμμίσω. Αυτά που κάνετε περιλαμβάνουν ορισμένα θετικά στοιχεία και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θα πρέπει από μαζί να τα εξετάσουμε για να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Σε αυτά τα οποία αναφέρει ο δικός σας χάρτης της 17ης Ιουνίου, από τα τέσσερα σενάρια διαλέξατε το δεύτερο σενάριο που είναι να βασιστείτε στον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση και την Προστασία από τις Χημικές Ουσίες για να καθορίσετε ποια είναι τα προϊόντα που έχουν ενδοκρινικά διαταρακτικό χαρακτήρα. Επομένως, η προσέγγιση σας δεν λαμβάνει υπόψη την, ε, τον ενεργητικότητα μιας ουσίας που χρησιμοποιείται σε, στη χημική βιομηχανία. Πολλοί από εμά επίσης λυπούμεθα γιατί δεν δεχτήκατε οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση των ουσιών. Να πείτε ότι είναι ενεργές ουσίες, είναι υποψη, ύποπτα για να είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, είναι σίγουρο ότι είναι διαταράκτες, όλο αυτό θα ήταν μια σημαντική πρόοδος. Και αυτό το πιστεύουν όπως ελέγχθη και οι ενδοκρινολόγοι. Γιατί ο δυνητικός κίνδυνος μιας ουσίας δεν μπορεί να ε, αποκλειστεί. Και αυτό που κάνετε στο σενάριο 2 δεν μπορείτε εσείς να ξεχάσετε ότι ορισμένες ουσίες έχουν ενδεχόμενο κίνδυνο να είναι διαταράκτες. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο 2013-2020 για την έρευνα, τότε η Κομισιόν είχε ε, δεσμευτεί να, παρουσιάσει οριζόντια κριτήρια για την κατάταξη των ενδοκρινικών διαταρακτών. Αυτό το οποίο παρουσιάσατε εσείς θα έπρεπε να καλύπτει όλες τις μορφές νομοθεσίας που εμπλέκουν τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. και υπάρχουν παντού γύρω μας στα καλλιντικά, στις συσκευασίες, στα παραστοκτόνα, ακόμα και σε ιατρικά σκευάσματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές πίεσεις που σίγουρα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το Σώμα των Επιτρόπων για τα θέματα αυτά. Πιστεύουμε όμως και λυπούμεθα για το γεγονός ότι η θέση της Κομισιόν δεν επεκράτησε έναντι των Επιτρόπων οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τον οικονομικό αντίκτυπο της σε βάθος κατάταξης παρά για τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε λοιπόν στην εξέταση αυτού του νομοθετικού πακέτου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο μακριά όπως εσείς θελήσατε στην αρχή. Στην ε, κατάταξη αυτή που θα επιτρέψει να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των πτυχών της ε, υγείας και της ε, προστασίας του περιβάλλοντος για του διαταράκτες. Ευχαριστώ. Η κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, τόσο σύντομα μετά από την χρεσινή παρουσίαση της πρότασης της Κομισιόν. Και επανέρχομαι στην χθεσινή διάσκεψη τύπου. Είπατε χθες ότι η Κομισιόν πήρε το δεύτερο σενάριο. Αυτό όμως δεν είναι σωστό απόλυτα, γιατί το δεύτερο αυτό σενάριο των ορισμών του Παγκοσμίου Οργανισμού ε, Υγείας περιλαμβάνει και την ανάγκη, δεν περιλαμβάνει την ανάγκη να αποδειχθεί η αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Εδώ αλλάζεται το βάρος της αποδείξεως. Εμείς πάντα είχαμε την αρχή της πρόληψης όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να αποδείξει κανείς ότι κάτι είναι αυλαβές και όχι να αποδείξει κανείς ότι είναι βλαβερό. Αυτό το οποίο κάνετε λοιπόν παραβιάζει τις αρχές της καλής νομοθεσίας που περιλαμβάνει και την αρχή της πρόληψης. Εγώ δέχομαι κριτήρια που βασίζονται σε επιστημονική γνώση. Αλλά αν δείτε την ε, αξιολόγηση του, της γλυφοσάτης από την ΕΦΣΑ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει καμία ε, επιστημονική γνωμοδότηση από αυτούς οι οποίοι καταδικάζουν την γλυφοσάτη. Και εσείς θέλετε να εμποδίζετε τις ε, επικίνδυνες ουσίες μόνο όταν υπάρχουν αποδεδειγμένες αρνητικές επιπτώσεις. Μα με τον τρόπο αυτό θα είναι πολύ λίγες οι ουσίες που θα απαγορεύσετε εσείς. Και επίσης, εσείς λαμβάνετε υπόψη τις εκθέσεις του παραγωγού αυτών των ουσιών. Και αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερα. Ε, μας ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι εσείς επί τρία χρόνια προετοιμάζετε μία απόφαση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη πραγματικά τα επιστημονικά κριτήρια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και ξέρω ότι δεν φταίτε εσείς προσωπικά. Δεν θέλω να ρίξω το φταίξιμο σε εσά. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Κομισιόν. Εδώ και ένα χρόνο τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή απόφαση για τα θέματα αυτά. Αλλά θα υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα πρόσφυγη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα αναγκαστούμε να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν από τρία χρόνια. Αυτό είναι μια μεγάλη απογοήτευση. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά έχουν ήδη υποθεί. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να περιοριστώ στα συγκεκριμένα ζητήματα. Χθες παρουσιάσατε μια πρόταση κυρίως για ζυζανιοκτώνα και βιοκτώνα. Μακροπρόθεσμα όμως αυτή η κολυσιεργία και επίσης αυτή η ταξινόμηση των ουσιών θα πρέπει να επεκταθεί σε άλλου τομεί. Σε το φορές διατάραξης και το ερώτημά μου είναι πότε μπορούμε να την περιμένουμε αυτή την επέκταση για να καλύπτει και συστατικά τροφίμων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ενδοκρινικοί διατάρακτε και στα τρόφιμα. Οι καταναλωτές πότε μπορούν λοιπόν να περιμένουν να ρυθμιστεί και αυτό για να είναι καλύτερη προστασία τους. Δεύτερο ερώτημα. Πρέπει κανείς να δείξει, αλλά και να αποδείξει ότι είναι επικίνδυνος ένα ενδοκρινικός διατάρακτης. Οι Δανείοι επιστήμονες έχουν κάνει πολύ καλούς υπολογισμούς και αξιολογήσεις ε, με βάση κλινικές δοκιμές σε ζώα, αλλά εξέτασαν και ε, τον άνθρωπο, φθόριο, φθόριουχα, Άρα ε, στα τρόφιμα μπορούν να οδηγήσουν σε αποβολές, για παράδειγμα. Μπορείτε να κάνετε έρευνα βέβαια σε αυτό και να πείτε ότι ακριβώς αυτή η συγκέντρωση αυτού, αυτής της ουσίας μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή. Όμως, αν κάτι θέλετε ότι είναι αποδεδειγμένο, η υπόθεση των επιστημόνων που δεν μπορούν όμως να προσδιορίσουν ακριβώς ε, το ποσό, την περιεκτικότητα, πώς θα αντιμετωπίζετε, δεν θα αντιλαμβάνετε υπόψη. Κύριε Στάς, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κύριε Επίτροπε και ήρθατε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Συμφωνώ με αυτό που είπαν οι προλαλήσαντες, αλλά έχω και εγώ να πω κάποια θετικά πρώτα απ' όλα. ιδιότητα Το άλλο το οποίο είναι πολυθετικό είναι ότι δεν βασίζεστε μονάχα σε οικονομικά κριτήρια, αλλά με εντυπωσιάζει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε πάντα να υπάρξει αυτή η προσέγγιση. Υπάρχει η οδηγία του Δεκεμβρίου 2014 που δεν σας επιτρέπει να έχετε κάποια άλλη αντιμετώπιση και επανέρχομαι σε αυτά που είπε η Ενδοκρινική Ένωση που είναι επιστήμονες υψηλού επίπεδου και είπαν ότι τα κριτήρια τα οποία προτείνετε εσείς δεν θα έχουν σε αποτέλεσμα να υπάρξει μια πραγματική προστασία της ανθρώπινης και ζωικής υγείας. Και ότι τα κριτήρια αυτά θα οδηγήσουν σε ρύθμιση και απαγόρευση ενδεχομένω ελαχίστων και μόνο ουσιών. Και υπάρχει και το θέμα του οικονομικού κόστους που θα προκύψει από την δράση αυτών των ενδοκρινικών ουσιών. Έχετε λοιπόν, είχατε τέσσερις ε, επιλογές για τη δράση. Εκεί υπήρξε κάποια αξιολόγηση για το πόσες είναι οι ουσίες, οι ενδοκρινικοί διατράκτες που θα καλυφθούν από τη ρυθμισή σας. Δεχτήκατε μια ε, επιλογή που λέτε ότι είναι επιλογή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει αρχικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Περνάτε από μία ε, προσέγγιση ενδεχομένου κινδύνου σε μία ε, προσέγγιση κινδύνου μονάχα αποδεδειγμένου. Αυτό όμως θα οδηγήσει στο να υπάρχουν ενδοκρινικοί διαταράκτες οι οποίες θα είναι ελάχιστοι που θα ρυθμίσουν. Πόσες ουσίες θα καλυφθούν λοιπόν από την δική σας ε, ρύθμιση αυτή τη στιγμή. Και επίσης αυτό το οποίο είπε ο Μπάς Ακάουτ. Το πέρασμα από το hazard στο risk, αυτό δεν συνάδει με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής. Δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό με το να τροποποιήσετε με τον τρόπο αυτό την βασική νομοθεσία. Πώς θέλετε να αντιδράσετε λοιπόν σε αυτές τις επικρίσεις. Ευχαριστώ. Κύριος Καπούτο, τελευταίο θα λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Μόλις 24 ώρες αφού πέρασε αυτό το μέτρο όπως είχατε πει μας τα προσφέρετε πριν τις ε, διακοπές, προβληματίζουμε σχέση με αυτό που αποφασίστηκε. Όχι μόνο εγκρίνατε αυτόν τον πάρα πολύ στενό ορισμό σε σχέση με τους διαταράκτε, το τι είναι δηλαδή διαταράκτε, αλλά έχετε τώρα και κάποιες ευρύτατες εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις. Έχουμε τον ορισμό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Οπότε εδώ πέρα προκύπτουν κάποιες διαφορές. Τονίζετε εσείς το ότι χρειάζεται να αποδειχθεί ότι υπάρχει κάποια αιτιώδης σχέση μεταξύ των αρνητικών επιδράσεων επί της ε, υγείας και ε, του διατάρακτη. Και είπατε ότι ε, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από κάποια πειράματα που όμως δεν είναι τόσο, τόσο στέρεα, τόσο στεγανά αυτά τα Οπότε η ουσία αυτή αλλάζει τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος. Όμως, κάποιες ουσίες θα απαγορευθούν και είπατε ότι αυτές θα είναι το πολύ 26. Όμως, ο έχει αμφισβητήσει 800 τέτοιες ουσίες. Θα πρέπει νομίζω να μας διευκρινίσετε κάποια πράγματα τα οποία είπατε στην εισήγησή σας, γιατί ανησυχούμε και ακόμη περισσότερο για την ισχύουσα νομοθεσία. Είπατε ότι αυτές οι ουσίες είναι ουσίες οι οποίες δύναται να δημιουργήσουν αρνητικά βλαβερά αποτελέσματα. Και αν υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργήσουν κίνδυνο. Υπάρχει όμως και το θέμα της έκθεσης σε κίνδυνο, είπατε. Τι γίνεται με τα παρασιτοκτόνα, Νομίζω ότι πέρα έχουμε μια φαιά ζώνη εκεί όπου ε, ασκείται σαν μου σα. Μα ξέρουμε τι έγινε και με τη γλυφοσάτη. Θέλετε να συνενέσουμε ούτως ώστε να γίνει η Ευρώπη πρωτοπόρα σε αυτό το μέτωπο. Ε, κύριε Επίτροπε, δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είστε πιο φιλόδοξοι ως Επιτροπή σε σχέση με την ε, αρχή της προφύλαξης να την εφαρμόζετε και να έχετε επίσης υπόψη το ότι εμείς το πρώτη μας προτεραιότητα που έχουμε είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και όχι τα οικονομικά επιχειρήματα. Ο Πρόεδρος, ε, εμείς σας ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος για να απαντήσει. Ευχαριστώ συνάδελφε. Είμαι ευχαριστημένος, είμαι καταχαρούμενος γιατί αποδείχθηκε ότι είμαστε στη σωστή ρότα. Σε έναν δεν αρέσει το ένα, σε άλλο δεν αρέσει το άλλο, στον τρίτο κάτι άλλο παραπέρα. Κύριε Χάζεκαμπ, είπε ότι δεν θα πρέπει να παίζουμε με την υγεία του κόσμου. Εγώ δεν είμαι ο δόκτωρ Μέγκελε. Είμαι ο δόκτωρ Κάιδες και ουδέποτε έχω παίξει με την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλώ μη λέτε τέτοια πράγματα. Γιατί, γιατί, με τίποτα, με τίποτα δεν είναι δυνατόν να συζητούμε τέτοια θέματα ηθικής ε, απόχρωσης. Σας ξαναλέω, δεν είμαι ο Μέγκελε. Ναι, είμαι γιατρός και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να έχουμε κάποιο είδου ε, διάγνωση κλινική. Υπάρχουν ε, διαφοροποίησει, αποχρώσεις. Μου είπατε για την εταιρεία των ε, ενδοκρινολόγων. Έχουμε δηλώσεις επιστημόνων. Ωραία, έχει την άποψή τη και σεβαστή η εταιρεία ενδοκρινολόγων. Αλλά έχει άλλη άποψη η εταιρεία τοξικολογίας. Και αυτή είναι σεβαστή. Όμως, η νομική πλευρά του θέματος ε, είναι κάτι που δεν ξέρω εγώ, αλλά ούτε και εσείς. Στην προηγούμενη θητεία είχαν γίνει τέτοιου είδους ε, κρίσεις νομικού επίπεδου. Επισήμανση κινδύνου, αξιολόγηση κινδύνου κλπ. Το ίδιο για το χάζατο όπως και για το ρίσκ. Κίνδυνος και διακινδύνευση ας πούμε αλλά και εσείς και εμείς στην Επιτροπή διαχειριζόμαστε το κίνδυνο και τη διακινδύνευση. Δεν παίζουμε. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε στο ίδιο γήπεδο. Έχουμε τρία επίπεδα, είπαμε, για να το διαχειριστούμε. Πρώτα-πρώτα την Επιτροπή, μετά περνάμε στο Κοινοβούλιο και μετά στα κράτη-μέλη. Άρα θα πρέπει έτσι να τα βλέπουμε συνολικά τα πράγματα και να δούμε το πώς μαζί, χέρι-χέρι θα προχωρήσουμε. Να μην παίζουμε με το τι λέει ο ένας φορέας και τι λέει ο άλλος. Υπάρχουν ενδείξεις για το ότι υπάρχει αβεβαιότητα και διάσταση απόψεων των επιστημόνων. Γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να ανασυστήσουμε τα αποτελέσματα τέλο πάντων. Υπάρχει προβληματική ακόμα. Είναι απίθανο στο εγγύς μέλλον να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι επιστήμονες. Μιλάμε για 23 εξέχοντες επιστήμονες που προσυπέραψαν αυτό το οποίο σας είπα. Μην κολλάτε μόνο σε μία πηγή. Πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει αβεβαιότητα για αυτό το τόσο δύσκολο θέμα. Και η απόκληση των απόψεων δεν αφορά μόνο την επισήμανση του κινδύνου. Υπάρχουν και διαφορές στη μεθοδολογία. στο τι μέσα θα χρησιμοποιήσει η έρευνα είναι δύσκολο, περίπλοκα τα θέματα. Για να δούμε τώρα. Ξεκινούμε από την κυρία Γκροστέτ. Μας είπε και αυτή την ε, προσέγγιση επί τη βάση του Χάζελ. Δεν έχει αλλάξει αυτό που θέσπισε ο κανονισμός. Έχουμε τους δύο σχετικούς κανονισμούς και αν μια ουσία χαρακτηριστεί ως διαταράχης, τότε θα απαγορευτεί. Εκτός εάν ισχύει κάποια εξαίρεση, παρέκκληση. Είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι επιστημονικές ε, ενδείξεις το πόσο δυνατή είναι η ουσία, το πόσο κίνδυνο ε, ενέχει κλπ. κλπ η έκθεση δεν αρκεί σαν κριτήριο. Χρειάζεται μια πλήρης αξιολόγηση του κινδύνου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επικαιροποιήσει τις παρεκκλήσεις για τα ε, παρασύτοκτονα. Και όταν επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παρέκκληση θα πρέπει να ενημερώνει σχετικώς. Είπαμε για αυτή την δήλωση των 20 τόσων επιστημόνων και είπαμε ότι η ισχύ statement also that... Λοιπόν, είπαμε ότι έτσι θα πρέπει να γίνεται από τη βάση του κινδύνου και όχι μόνο της δραστικότητας, potency. Αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Είναι πολύ περίπλοκο. διάφορες κατηγορίες. Κατηγοριοποίηση δεν μας οδηγεί σε βελτίωση του ορισμού. Το ίσως δεν σημαίνει σίγουρα. Εμείς ως ε, νομοθετική εξουσία θα πρέπει να δρούμε άμεσα. Η κατηγοριοποίηση δεν ωφελεί στην υγεία και στο περιβάλλον. Το μόνο το οποίο κάνει είναι να δημιουργεί μια φαιά περιοχή, μια γκρίζα ζώνη και δεν υπάρχει έτσι ασφάλεια κινδύνου ούτε για τις αρχές ούτε για τους ε, εμπλεκομένους. Γιατί είπαμε ποιες είναι οι συνέπειες για τις διάφορες κατηγορίες και για τα βιοκτώνα και για τα παριστοκτώνα και για την ομοδασία που τα διέπει. Αναφέρατε ορισμένοι ξημών ότι είναι ζητήματα οριζόντια. Ωραία, όλοι προβληματιζόμαστε. Πώς θα προχωρήσουμε. Έχουμε το Ρίτσα, έχουμε τα καλλιντικά, έχουμε τα είδη διατροφής, την οδηγία για το νερό. Πολλά νομοθετήματα υπάρχουν. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Αυτό δεν είναι ζήτημα μόνο του σήμερα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κριτήρια για τους διαταράκτες και μετά δούμε πώς θα χειριστούμε την ε, νομοθεσία και τον κανονισμό για βιοκτώνα και παραστοκτώνα. Αυτή είναι η εντολή μου σήμερα. Ωραία, εάν μπορέσουμε θα προχωρήσουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Και εμένα μου φάνηκε παράδοξο. Γιατί έχουμε αυτού του διαγωνισμού παρεστοκτών και διοκτώνα και είπαμε ότι αν έχουμε έναν ε, διαταράκτη με βάση αυτών θα απογραφτούν. Αν όμω ε, είναι κάτι που σχετίζεται με τα τρόφιμα, ισχύει άλλο νομοθέτημα. Μα δεν καταλαβαίνω. Άρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό είναι το βήμα που θέλω να κάνω. Αυτό είναι η δουλειά μου σήμερα. Να βρω κάποια κριτήρια σύμφωνα με την ε, εντολή που έχω με τους δύο αυτούς κανονισμούς. Και σήμερα με τον κανονισμό ε, της προστασίας και βέβαια θα πρέπει να συζητήσουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Επίσης, Μπάρτ. Μπάς, μπάς. Ο μπάς Έκχαλ. Ακόμα δεν έχουμε εντοπίσει κάποιες ε, ουσίες που έχουν ιδιότητες διαταράκτη. Μιλάμε για 347 ουσίες που εξετάστηκαν. 25 χημικές ουσίες αναφέρθηκαν ως διαταράκτες. 25 ουσίες. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας πλήρους αξιολόγησης, αλλά αυτό μας δίνει να καταλάβουμε το, την τάξη μεγέθους για το τι αξιολόγηση πρέπει να γίνει. Οπότε θα πρέπει η ΕΦΣΑ να επιληφθεί. Στο μέλλον όμως βεβαίως θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της ε, επιφύλαξης και προφύλαξης στο επόμενο βήμα. Μιλάμε για τις πιθανότητες και άρα θα πρέπει η αρχή της προφύλαξης να εφαρμοστεί με τον πιο σωστό τρόπο και να είμαστε προσεκτικοί όταν παρεμβαίνουμε σε αυτή την κατάσταση. Ε, ο Μπάσεκ Χαβγε το πήραμε τα μεταζώα. Η αξιολόγηση για τις χημικές ουσίες όσον αφορά τις ενδεχόμενες ιδιότητες διαταρακτών ε, σημαίνει ότι υπάρχουν τοξικολογικά δεδομένα αντίστοιχα τα οποία βγαίνουν από μελέτες και πειράματα με τα ζώα. Αυτό ήδη γίνεται σε επίπεδο ΩΣΑ και από την υπηρεσία την αντίστοιχη των ΙΠΑ και είπαμε ότι θα κάνουμε το επόμενο βήμα προς την τοξικολογία στα, σταματώντας τα πειράματα με τα ζώα. Και κατά θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που η νομοθεσία καλύπτει τους διαταράκτες με σκοπό την στεγανή προστασία και τη ρύθμιση για τα βιοκτώνα με ξεκάθαρα κριτήρια επί τη βάση μιας σύγχρονης επιστημονικής προσέγγισης. Μόνο τα αρνητικά αποτελέσματα των ουσιών ελήφθησαν υπόψη από τον νομοθέτη. Και έτσι μπορούσαμε να λάβουμε τη σωστή απόφαση σε σχέση με την απαγόρευση κάποιων ουσιών. Για μένα ήταν πολύ δημιουργική αυτή η συζήτηση. Και θα ξαναδιαβάσω αυτά τα οποία ρωτήσατε και θα σας απαντήσω συμπληρωματικά. Είπαμε, πολύ μου αρέσει η σημερινή ζήτηση γιατί του ενός δεν του αρέσει το ένα, του άλλου δεν του αρέσει κάτι άλλο. Αυτό πάνω να ότι λάβαμε τη σωστή απόφαση. Σας ευχαριστώ. Ακούστε. I am in, Green Party. I am in, in, I see all, all uh, colors in Δεν είμαι πράσινος, λέει ο κ. Τα βλέπω όλα τα χρώματα εδώ. Είναι πολιτικό, δεν είναι πολιτικό. Λοιπόν, ε, ο Πρόεδρος, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση επί του σημείου αυτού. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο που ήρθε. Ακούσαμε κάποιες απαντήσεις, ίσως όχι όλες που θέλαμε να ακούσουμε αλλά θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Και βέβαια, εφόσον το επιθυμούμε, έχουμε και τη δυνατότητα να προσβάλλουμε αυτή την πρόταση, να υποβάλουμε ένσταση κατά της πρότασης αυτής. Okay, dear colleagues. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει περάσει η ώρα. Αλλά μπορούμε να περάσουμε ευθύ αμέσω στο επόμενο σημείο τη μερίσια διάταξη. Που είναι η βασική στόχη για τη 17η Σύνοδο τη ΣΥΤΕ. Συμβαλωμένο μερών τη ΣΥΤΕ. Έχουμε ψηφίσματος ψηφίσματο. εκ μέρου του ΕΛΚ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται τώρα για την ΣΥΤΕΣ ή ΣΑΙΤΕΣ, την συμφωνία αυτή, η οποία είναι μεγαλύτερη συμφωνία μέχρι στιγμή για την προστασία των απειλουμένων φυτών και ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν μεγάλες ευκαιρίες να λύσουμε το πρόβλημα αυτό με ένα βιώσιμο τρόπο και να αποτρέψουμε την παράνομη θηρία, την παράνομη θύρα των ζώων. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να συζητήσετε για το προηγούμενο θέμα, κάντε το έξω παρακαλώ, λέει ο Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μα και ξαναδίνω στον κύριο Λίνη το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε πρόεδρε. Κάθε τρία χρόνια γίνεται μια συνδιάσκεψη των συμβαλωμένων κρατών εφέτος θα γίνει στο Johannesburg το Σεπτέμβριο <clears throat> γιατί συζητούμε για το θέμα αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται για πρώτη φορά αφού προσυπέραψε το 2015 στην συνδιάσκεψη αυτή. Το εμπόριο για απειλούμενα είδη είναι μία από τις πιο κερδοφόρες μορφές εγκληματικότητος και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει από κοινού να το αντιμετωπίσουμε. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το παράνομο αυτό εμπόριο με κυρίως τη ζήτηση της ζήτησης. Η Ευρώπη είναι πολλές φορές η τελικός προορισμός ή ο χώρος διαμετωκόμησης αυτών των προϊόντων και επομένω παίζει κομβικό ρόλο. Χαίρομαι για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κομισιόν το Φεβρουάριο προ... έτεινε ένα σχέδιο δράσης και τώρα εμείς πρέπει να παρουσιάσουμε μια έκθεση πρωτοβουλία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και αυτό έχει και σημαντικό ρόλο για την συνολική αυτή δράση για τα προστασία των απειλουμένων ειδών. Και θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την υποστήριξή τη στην διάσκεψη ΣΥΤΕΣ και από την πλευρά του Συμβουλίου υπήρξε μια θετική ανταπόκριση. Την επόμενη Δευτέρα θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εγκληματικότητα που συνδέεται με τα άγρια είδη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Προεδρία της, ε, των κάτω χωρών και επίσης και η επερχόμενη Προεδρία της Σλοβακίας έχει παίξει έντονο ρόλο στα θέματα αυτά. Εμείς έχουμε μια σειρά από ερωτήματα που συμφωνήσαμε να θέσουμε στην Κομισιόν για την στοχοθεσία που θα ακολουθήσει η Κομισιόν και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στη, στην ε, συνδιάσκεψη αυτή και θα έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος που να περιλαμβάνει τις ε, τα αιτήματά μας και τις προτάσεις μας για την Κομισιόν στην διασκευή του που αυτό το οποίο ακόμα δεν βρίσκεται στο ε, ψήφισμα, είναι το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την συνέχιση της θύρας με έναν τρόπο ο οποίος όμως να είναι βιώσιμος και να καλύψει και τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται στις περιοχές που υπάρχουν άγρια ήδη υπάρχουν τώρα οι δυνατότητες από τους συναδέλφους να θέσουν τροπολογίες μέχρι την επόμενη Τρίτη για τα θέματα αυτά. Περιμένω λοιπόν, θέλω να ε, χαιρετήσω και τις προτάσεις Κομισιόν για την αντιμετώπιση της παράνομης ε, θύρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για μένα γιατί είναι ένας κίνδυνος για την ε, βιοποικιλότητα και την αηφόρο ανάπτυξη αλλά και για τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων στις χώρες όπου βρίσκονται αυτά τα είδη. Πρέπει η οργανωμένη εγκληματικότητα, η οποία χρηματοδοτείται από τέτοιες ε, δραστηριότητες να κατασταλεί και να δοθεί στους ανθρώπους εκεί να μπορούν να ζήσουν και να ε, βρίσκονται σε συνθήκες οι οποίες θα είναι ομαλές και συνθήκες ευμάρειες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την αρισίδα εγκλήματος να υπάρξει δίωξη και συμμετοχή όλων των αστυνομικών αρχών, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από τις υπόλοιπε χώρες του κόσμου, να υπάρξει απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοκτικών <clears throat> αρχών και εδώ εμπλέκεται προφανώς η Europol, η Interpol, η Eurojust και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν να δώσουν ένα πολύ καλό παράδειγμα με τη συνεργασία στον τομέα αυτό. Αναφερόμαστε επίσης και στο ψήφισμα στα είδη που πρέπει να καλυφθούν από, το, από την συμφωνία αυτή. Εγώ θα ήθελα να έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα συγκεκριμένα είδη όπως είναι ο Αφρικανικός ελέφας ή ο Αφρικανικός λέων ή ο Λευκός ρινόκερος, είδη τα οποία χρήσουν προστασίες. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε πια αυτά τα είδη και να δώσουμε έτσι ένα σαφές μήνυμα. Συγγνώμη και σας ζητώ συγγνώμη γιατί θα πρέπει να φύγω σε λίγο γιατί έχω μια σημαντική συνάντηση. Σας ευχαριστούμε Παύλ Πότς, Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και το συνάδελφό μου για να μην δαπανίσουμε πολύ χρόνο, να πω ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία οι συνεισηγητές. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία και τους εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν όλα τα ε, υλικά και όλη την τεκμηρίωση. Νομίζω ότι είναι καλές προτάσεις, τη στηρίζει η ομάδα μου, όπως και τη δέσμευση και το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας. Υπάρχει το σχέδιο ψηφίσματος, όμως για τα παραρτήματα δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες, δεν συμπεριληφθεί η πρώτη ε, στην κατάρτιση του πρώτου ε, προσχεδίου. Θα κατατεθούν πάντως τροπολογίες ε, από τους συνεισηγητές. Έχουμε με τεχνική συνεδρίαση αργότερα για το παράνομο κυνήγι. Σίγουρα είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Θα καταθέσω και άλλες τροπολογίες. Είναι πλοκό πάντως το θέμα. Περιμένω λοιπόν να έχουμε ένα καλό συντονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μαρή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τους συνεισηγητές, να τους ευχαριστήσω. Ήταν εξαιρετική η δουλειά που κάναμε, πιστεύω. Έχουμε φτάσει σε αυτό το κοινό ψήφισμα που προτείνει νομίζω μια φιλόδοξη θέση για την επόμενη διάσκεψη των συμβαλωμένων μέρων. Θα ήθελα επίση να απογραμμίσω έναν πολύ καθοριστικό ρόλο που έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα. Πιστεύω ότι είναι εφικτό σε αφορά την προστασία της βιοπικιλότητα. να είμαστε ε, το ίδιο ε, διορατικοί και προβλεπτικοί και να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το κυνήγι τροπέων ε, θα καταθέσουμε τροπολογίες γιατί τη δραστηριότητα αυτή θεωρούμε ότι είναι επαρχιωμένη και πρέπει να το υπενθυμίσουμε ότι είναι και κληρονομιά από την αποικιοκρατική εποχή. Θα πρέπει νομίζω να προβληματιστούμε για μια αναδιατύπωση ε, μάλλον για μια αναμόρφωση των σχέσεων του ανθρώπινου είδους με το άλλα ε, έμβια όντα. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αποκεντρωσμένες πρακτικές. Έχουμε τεράστια ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μία από τις σημαντικότερες αγορές μετακόμισης και εισαγωγής και δεν μπορούμε να υπολοιπόμεθα ε, των ε, προσπαθειών που πρέπει να γίνουν για αλλαγή νοοτροπίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Τέιλορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πράσινοι είμαστε ικανοποιημένοι με το σχέδιο ψηφίσματος και για την ε, αρμονική προσέγγιση των συνεισυχητών μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Από ό,τι φαίνεται θα συμφωνήσουμε όλοι όχι μόνο για τη ζωτική σημασία της 17ης διάσκεψης των συμβολωμένων μερών τη ΣΥΤΕΣ για την προστασία ε, των ειδών άγρια πανίδα σε διεθνέ επίπεδο, αλλά σίγουρα και η Ένωση μπορεί να συμβάλλει ζωτικά για τη βελτίωση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και τις δομές τις σχετικές και να είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της μαζικής διαφθοράς που έχουν στα εμπόρια των Αγρία πανίδας. Αναγνωρίζω ότι η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλον έχει ήδη κάνει αρκετά για να μειώσει και το κίνδυνο από το κυνήγι τροπέων και να επιβάλλει πιο αυστηρά ε, περιορισμούς ε, για το κυνήγι των ειδών του παρατήματο 1 και 2 της ΉΤΕΣ. Επίσης αναγνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει και ένα ρόλο και μπορεί να απευθύνει έκκληση και σε άλλους συμβαλωμένους στις σάιτες για να εγκρίνουν αυτή την πρόταση. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένα είδη πανίδας, εγώ είμαι υπέρ της εφαρμής αρχής προφύλαξης. Έχω διαβάσει πολλές από τις προτάσεις για την προστασία ειδών όπως ο Αφρικανός ελέφαντος, λευκός, ε, ε, ρινόκερος, ε, η τίγρης, οι αφρικανικοί λέοντες και άλλα ελουροειδή. Η Ένωση πρέπει να τα στηρίξει όλα αυτά. Υπάρχουν και πολλά ήδη αφρικανικά και ασιατικά που έπρεπε να πάνε στο παράρτημα 1. Γιατί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 Πολύ χρήσιμη ήταν η συνάντηση στο Στασβούργο με τους ειδικού κατά την τελευταία ολομέλεια. Μας βοήθησαν πολύ να κατε, καταλάβουμε τα τεχνοκρατικά, τεχνικά σημεία. Βέβαια, ε, ε, το θέμα εδώ είναι, έρχεται σε συνέχεια προηγούμενου προβληματισμού μας Τώρα είπαμε, τώρα θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά εδώ τα είδη, τα άγρια είδη. Και θα πρέπει επίσης να δονήσουμε ότι έχουμε 80.000 είδη ε, που, από τα οποία 23.000 λέει ο ΙΕ κινδυνεύουν από εξαφάνιση. Είπαμε ότι είναι θέμα διαφθοράς και έτσι γίνεται αυτό το παράνομο εμπόριο. Θα πρέπει όμως να διατεθούν για την καταπολέμηση αυτού του λαθρεμπορίου ειδικοί πόροι. Εκεί στο τελευταίο τμήμα που αναφέρονται κάποια είδη έχουμε αυτές τις ε, τροπολογίες. Συμφωνούμε σε αυτές. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνει προσέγγιση ε, προφύλαξης. Και επί των δύο παρατημάτων θα πρέπει να βελτιώσουμε την διαδικασία πριν κάνουμε την ε, τροποποίηση του κειμένου. Να υπάρχει δηλαδή 100% επιστημονική βεβαιότητα σε σχέση με την απειλή εις βάρος αυτών των ειδών. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Ντορνάνο. Εδώ έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις εν ώψη της σύντησης του ΣΥΤ για ε, την απειλή εις βάρος κάποιων ειδών, χλωρίδας και πανίδας. Για πρώτη φορά ε, προβληματίζεται για αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για αυτό το λαθρεμπόριο και χρειάζεται επομένως μια προσέγγιση για την ανιχνευσιμότητα και την ευαισθητοποίηση. Αυτά νομίζω ότι είναι ό,τι χρειάζεται όσον αφορά το σημερινό πρόβλημα. Πάντως, πριν ενθουσιαστούμε για αυτή την προσέγγιση της Ένωσης για την ΣΥΤΕΣ, θα πρέπει να δούμε εάν τώρα υπάρχει μια πραγματική προσθεμένη αξία θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να αναβαθμιστεί ε, η, η, η, αποτελεσματικότητα της ΣΥΤΕΣ. Τι θε, μήπως τυχόν απειλείται η κυριαρχία των κρατών μελών μια που μιλάει εξ ονόματός της Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να δούμε ότι έτσι ε, ε, δεν θα πρέπει να αποκλείονται τα κράτη-μέλη από το να προσχωρήσουν ώστε άφτασε σε αυτή την σύμβαση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από κράτη έθνη ή έθνη κράτη. Υπάρχει όμω εδώ ένα παράδοξο. Τώρα όσον αφορά τη διαφάνεια της χρηματοδότησης και της ε, συγκρούσεις συμφερόντων αλλά και ε, την αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων εδώ πέρα υπάρχουν πολλά θέματα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν τώρα. Κύριο Σάντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την υποστήριξη που πήρα από ένα αριθμό εντύμων βουλευτών. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου στην συνδιάσκεψη των συμβαλωμένων μερών στο Johannesburg. Χαιρετίζουμε λοιπόν το ψήφισμά σας, όπως ελέγχθη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική συνδιάσκεψη. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει ως ε, συμβαλόμενο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσθέσει αξία. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ως Βρετανός τώρα πρέπει να είμαι <laughs> προσεκτικός όταν λέω ότι είμαστε όλοι ενωμένοι. Σίγουρα θα είναι σημαντικό το θέμα αυτό και έχουμε πολύ φιλόδοξες προτάσεις για αυτήν τη συνάντηση. Το θέμα είναι και κατά πόσο θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια ευρύτερη επιρροή. Προσπαθούμε να αποκομίσουμε στο δεύτερο περισσότερη υποστήριξη για τις προτάσεις μας. Αυτό τονίστηκε στην πρόσφατη συνάντηση της Ναϊρόμπη του υπηρεσιών του ΟΗΕ και στους G7 υπάρχουν διάφορα διαβήματα που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες του κόσμου με στόχο να φέρουμε την προσοχή τους στις προτάσεις μας και να τις υποστηρίξουμε. Βλέπουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησή σα και χαιρόμαστε για το γεγονό ότι υποστηρίζει ιδιαίτερα το έργο τη Κομισιόν. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει σύγκρουση και διαφορά μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν αναπτυχθεί μέσα στα πλαίσια της ε, Σύμβασης Σάιτες και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει θετική απόλυξη στο Συμβούλιο την ε, ε, Δευτέρα στο Συμβούλιο και φυσικά και η Ολλανδική Προεδρία θα πρέπει να σας πει γι' αυτό. Θέσατε ορισμένα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, το θέμα της διαφάνειας και της λειτουργίας της Σύμβασης ΣΑΙΤΕΣ. αυτό είναι ένας τομέας όπου εμείς έχουμε προτείνει ένα ψήσιμο το οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά και θέλουμε να γίνουμε πιο σαφή τρόπο στην πράξη. Υπήρξαν επίσης θέματα που αναφέρθηκαν για την τροπεοθυρία και εδώ προτείνουμε οι σάιτες να ενισχύσει τα θέματα για την θύρα τροπέων. Ε, άκουσα να αναφέρονται συγκεκριμένα ορισμένα είδη. Η προτάση μας, αφορά ένα ευρύ φάσμα ε, ειδών που θέλουμε να ενισχύσουμε με τη σύμβαση σάιτες στην προστασία τους. Πιστεύω λοιπόν θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική συνάντηση. Εμείς θα είμαστε ιδιαίτερα ε, παρόντες, θα είναι παρόν ο Επίτροπος Βέλα στις πιο σημαντικές συναντήσεις της συνδιάσκεψης και με τον τρόπο αυτό θα υπογραμμίσουμε την πολιτική και τεχνική σημασία αυτής της σύμβασης και την προσήλωση σε αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 21 Ιουνίου το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα είναι στις 12 Ιουλίου και θα πάμε στο Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημέρας διαταξής μας. Ανταλλαγή με απόψεων με την Ολλανδική Προεδρία για το νέο σχέδιο δράσης εναντίον της λαθρεπορίας αγρίων ειδών και έχουμε εδώ την Ολλανδική Προεδρία, στην οποία θα δώσω αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο της Ολλανδικής Προεδρίας, τον κύριο Λαμπεντέκερ, ο οποίος είναι αρμόδιος τα θέματα αυτά, για να κάνει τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις και μπορούμε στη συνέχεια να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ισότιμοι βουλευτέ τη Επιτροπή ΕΜΦΗ, είναι τιμή που βρίσκομαι εδώ για να ανταλλάξουμε απόψει ε, εκ μέρου τη Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το σημαντικό θέμα. Όπω όλοι γνωρίζουμε, το λαθρεμπόριο υγρών, ε, ειδών αγριάς πανίδας είναι πολύ ε, αποδοτικό και τροφοδοτεί την ε, ε διαφθορά, δωροδοκεί κυβερνήσει. Πολλές φορές ε, τις σειράξεις και την τρομοκρατία επηρεάζει αρνητικά τη βιοπικιλότητα, την άγρια ζωή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εκρίζωση της φτώχειας. Είναι ένα θέμα που επηρεάζει πολλούς τομείς, εγκάρσιο και δεν γνωρίζει σύνορα. Και δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο μακριά σε άλλε υπήρου. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αγορά σε διαμετακόμισης και πολλέ φορέ και προορισμού. Και έχει σίγουρα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Όμω δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση ε, Τώρα αρχίζει κάπως να βελτιώνεται η κατάσταση. Η, Γενική Διεύθυνση του ΟΗΕ, Περιβαλλοντική Συνέλευση και πέρυσι η G7 ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, αλλά και εσείς και η Επιτροπή σας όλους ιδιαίτερως ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα, όπως δείχνει το ψήφισμα που συζητήσατε πριν και η ημερήσια διάταξη σήμερα. Γνωρίζουμε ότι γίνονται πράγματα, κύριε Πρόεδρε, σε διάφορα κράτη-μέλη, από τι εθνικέ κυβερνήσει, όπω για παράδειγμα ε, στη χώρα μου η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει όλε τι ε, άδειε ε, για τρόπεοθυρία. Επειδή όμω υπάρχει αυτή ο διασαρκό χαρακτήρα, τα εθνικά μέτρα δεν αρκούν. Θα πρέπει να το δούμε διεθνώ το πρόβλημα. Η Ολλανδική Προεδρία λοιπόν έχει δώσει μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα αυτό και οργανώνουμε συνεδρίαση με το Act Now or Game Over. Η Κομισιόν ε, <coughs> παρουσίασε το σχέδιο δράσης ε, για την εμπορία, των, ε, την παράνομη εμπορία άγριας πανίδας. Μιλήσαμε για τη διατήρηση των ειδών, την συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης, των τελείων κτλ. Και με τις συζητήσεις αυτές ε, διατυπώσαμε μια αντίδραση σε αυτό το σχέδιο δράση από πλευρά Συμβουλίου. Θα περιλαμβάνεται και στα πορίσματα, στα συμπεράσματα που θα εγκρίνει στις 20 ε, Ιουνίου τη Δευτέρα δηλαδή το Συμβούλιο. Να σας πω ποιες είναι οι προσδοκίες μας, τι αναμένουμε από αυτή την συνάντηση. Νομίζω ότι θα εκφράσουμε την βαθιά ανησυχία μας για το θέμα του λαθρεμπορίου αγριάς πανίδας. Θα καλωσορίσουμε το σχέδιο δράσης ως σημαντικό μέσο για την αναβάθμιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση των εγκλημάτων σε όλα τα επίπεδα. όσο ό,τι φορά το λαθρεμπόριο Αγρίας θα ζητήσουμε όλοι να κάνουν ε, το, αυτό που του αναλογεί για το λαθρεμπόριο που πρέπει να σταματήσει. Και γι' αυτό απαιτείται καλύτερη συνεργασία μεταξύ ε, των αρχών επιβολής του νόμου, καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, απέλτιση των πρακτικών, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και κατάρτιση για τα όργανα επιβολής νομοθεσίας. Επίσης θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε ε, και μάλλον να ασχοληθούμε και με το διαδίκτυο Αυτά νομίζω θα εγκριθούν ε, τη Δευτέρα κύριε Πρόεδρε. Νομίζω είναι σαφές ότι είμαστε έτοιμοι ως Συμβούλιο να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να λάβουν δράση στο πλευρό της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου. Περιμένουμε λοιπόν την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και θα λάβουν τις απαιτούμενες αποφάσεις για να είναι αποτελεσματική κοινή μα προσπάθεια. Εδώ ολοκληρώνω την παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ. Thank you for the introduction. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισαγωγή. Μπορούμε να περάσουμε απευθεία στη συζήτηση. Το λόγο λοιπόν, συνάδελφος Ντορνανό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο με σάιτες από τις 8 Ιουλίου του 2015. Θα περιμέναμε λοιπόν το σχέδιο δράσης για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα να αποσκοπεί κυρίως στη στήριξη και την ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα αυτής της σύμβασης. Το κείμενο αυτό λοιπόν που ισχύει από το 1975 είναι θεμέλιο της δράσης μας στον τομέα αυτό, όμως το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον άγρια παράδοση ε, προτείνει 32 τράσεις που είναι καλοπροαίρετες, ε, όμως ε, το πλαίσιο είναι άκρος ευρωπαϊκό. Άρα οι σάιτες και τα κράτη συμβαλόμενα διαχωρίζονται με ένα τείχος και όλες οι κανονιστικές διατάξεις έχουν ως κίνδυνο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής και της προθεσμίας Καθυστερημένη εφαρμογή λοιπόν. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς, ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη χρηματοδοτούμε προγράμματα προστασίας θαλάσσιων ειδών ελεφάντων και άλλων ειδών, αλλά δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για ε, χρήματα των φορολογουμένων. Εμείς, η Γαλλία, είμαστε ένας από τους καθαρούς ε, χρηματοδότες. Η προσχώρηση της Ένωσης στο site της δεν θα πρέπει να είναι ένα πρόσχημα για μια ακόμη φορά να καταπατήσουμε την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών, που και αυτά είναι συμβαλόμενα με τη site της. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Ξέρω πόσο η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και πόσο προστασία των απειλούμενων των ειδών είναι κατεπίγουσα ε, και γι' αυτό η κυρίαρχη δράση των κρατών μελών. Ε, θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι έχει θέση σε αυτό τον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου άγριας πανίδας. Kolegové, já nemůžu odolat pokušení, aby tady zazněla čeština, takže teď i česky. se... Σας παρακαλώ λοιπόν να μιλάτε πιο αργά και δίνω το λόγο στον κύριο Μαζέ. Κύριο Σομαρζέ, δεν που μου δώσατε το λόγο. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε την Ολλανδική Προεδρία για τη στράτευσή της υπέρ αυτού του θέματος και ε, ελπίζουμε ε, να αναπτύξει την ίδια δραστηριότητα η Σλοβακική Προεδρία. Είναι πολύ σημαντικό το έργο πρέπει να επιτελεστεί ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην συνειδητοποίηση. Ε, ε, άρα πρέπει να συνεχιστεί η επικοινωνική εκστρατεία. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Το, το 1992 στο Ρίο είχαμε δύο πρωτόκολλα. Ένα όσον αφορά την ε, αλλαγή του κλίματος και ένα επίσης για την προστασία της βιοπικιλότητας. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανεί είναι ότι μετά 24 χρόνια το πρωτόκολλο για την βιοπικιλότητα καθυστέρησε πάρα πολύ όσον αφορά την εφαρμογή. Και το ίδιο επίση και τα μέτρα κατά της απώλειας της βιοπικιλότητας. Επομένως βρεθήκαμε σε αυτή την τραγική θέση όταν δηλαδή έχουμε τώρα το έκτο κύμα κατά τον ειδών. Ε, είναι εξαφάνισή του από τότε που ξεκίνησε η ζωή στον πλανήτη. Οπότε έχουμε τώρα ορισμένα αγρία είδη τα οποία θα πρέπει να τα προστατεύσουμε και είναι αυτό το οποίο ε, ονομάζουμε λαθρεμπόρια. Αυτό φταίει. Πρόκειται επομένω για την παράνομη εμπορία αυτών των αγριών ειδών. Οπότε θα πρέπει να προβληματιστούμε τα είδη είναι άγρια ή διακρίνει αγριότητα αυτό το εμπόριο γιατί τα ίδια αυτά τα οποία ονομάζουμε άγρια δεν έχουν πρόθεση να σκοτώσουν ανθρώπους και μετά να στολίσουν κανέναν τείχο με το κεφάλι τους. Επομένως, η αγριότητα χαρακτηρίζει την ανθρωπότητα, οπότε εδώ θα πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα και έτσι να ξαναθυμηθούμε τον ανθρωπισμό μας που δεν τον έχουμε τώρα μέσα στο σύνολο των απόψεων του πολιτισμού μας. Ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, εισαγωγή σας. Έχω δύο ερωτήματα. και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απόψή σας για τα θέματα αυτά. Το πρώτο ερώτημα αφορά την ε, υποστήριξη στην Ευρώπη και στον ΟΗΕ για να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο νόμος Λέιση που θα επιτρέπει την προστασία, που θα υποχρεώνει την προστασία των αγρίων ειδών από τη χώρα όπου βρίσκονται. Αυτό υποστηρίχθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2016 και αναφέρεται και στην έκθεση για το έγκλημα κατά των αγρίων ειδών και σε άλλες ιστοσελίδες. Εν όψη αυτού, λόγω αυτής της ε, ομοφωνίας που υπάρχει, θεωρεί η Ολλανδική ε, Προεδρία ότι θα πρέπει να περιληφθεί αυτό στο σχέδιο δράσης σας. Και το δεύτερο θέμα αφορά την ε, εμπορία σε εξωτικά κατοικίδια ήδη. Πολλά εξωτικά είδη βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα και έχουν εισαχθεί παραβιάζοντας τον νόμο των χωρών τους και δεν υπάρχει αρκετή εναρμόνιση στα θέματα αυτά για τους κανονισμούς σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ε, ζώων και τα οικοσυστήματα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε θετικούς καταλόγους για τα άγρια είδη που να επιτρέπουν μόνο ορισμένα τέτοια ζώα να εισάγονται. Γιατί έτσι θα υπάρχει μια σαφήνεια και για τις διοκτικές αρχές και για τους ιδιοκτήτες και θα μειώσει και τη γραφειοκρατία για τις κυβερνήσεις και θα επιτρέψει προληπτικά μέτρα. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για τη δυνατότητα να υπάρξει ένας θετικός κατάλογος για τέτοια ζώα. Ευχαριστώ. Ο κ. Χερμπράντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ολλανδική Προεδρία για να μας πει ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Όταν ξεκίνησα αυτόν τον αγώνα κατά του εγκλήματος, της εγκληματικότητας για τα άγρια είδη, αυτό ήταν κάπως καινούριο. Εγώ παρουσίασα ένα σχέδιο δράσης, πήρα από μια πρωτοβουλία για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και έχουν γίνει κάποιες σημαντικές πρόοδοι. Τώρα έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο δράσης η Κομισιόν πράγματι επέτυχε το στόχο της, έκανε αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί να κάνει. Ξέρουμε όμως όλοι ότι τώρα να πρόκειται στα κράτη-μέλη γιατί οι περισσότερες αρμοδιότητες που έχουμε, που έχουν να κάνουν με τα τελωνία, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη, είναι ναι. εθνικές αρμοδιότητες ναι. και όχι ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό στάδιο στον αγώνα κατά της λαθρεμπορίας αγριών ειδών. Και γι' αυτό εγώ κάπως επικρίνω αυτό που είδα στα σχέδια του Συμβουλίου, στα σχέδια συμπερασμάτων του Συμβουλίου, ότι τονίζεται η έννοια της επικουρικότητας σε διάφορα άρθρα και βλέπω ότι τα κράτη-μέλη προσκαλούνται να κάνουν κάτι ή ενθαρρύνονται ή τους λέμε ότι θα πρέπει να σκεφτούν, ίσως να σκεφτούν κατεπηγόντως αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Αν δούμε στα σοβαρά τι λένε οι υπουργοί μας και οι κυβερνήσεις μας, τότε δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο να προσκαλέσουμε τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αποφασίσουμε σε επίπεδο Συμβουλίου να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. ότι θα ενισχύσουμε τη συνεργασία, θα ενισχύσουμε και την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό. Είναι κάτι το οποίο πολύ απλό. Η Europol θέλει να δώσει πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ε, λαθρεμπορία αγρίων ειδών. χρειάζεται εντολή από τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται να υπάρξει και κάποια γραμμή, κάποια πρόταση στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που να ζητούν να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της λαθεμπορίας αγρίων ειδών. Δεν έχουμε πετύχει λοιπόν ακόμα το στόχο μας και εγώ φοβάμαι ότι το, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, αυτήν η φίλη μας που θα πρέπει να νοιάζονται για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να τεθούν όλα αυτά στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εμπορίου, εξωτερικών υποθέσεων, εσωτερικών και δικαιοσύνης. Θα το κάνει αυτό η Προεδρία και κατά πόσο θα ζητήσει να υπάρχουν στεναρά συμπεράσματα. Από ό,τι κατάλαβα, το αρχικό κείμενο, το οποίο εξετάστηκε στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου το Μάτιο, δεν αντιμετωπίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από τα κράτη-μέλη, αλλά τώρα έχει αλλάξει τα σχέδια συμπερασμάτων που έχω δει από το Συμβούλιο είναι υπερβολικά αποδυναμωμένα για να πάρει κανείς μια τέτοια πολιτική δηλωσή σοβαρά. Θα ήθελα να ε, ζητήσω λοιπόν να παροτρύνω την Ολλανδική Προεδρία να πάρει πιο σοβαρά το θέμα της ε, καταπολέμησης λαθρεμπορίας και όχι μονάχα να λέει ότι προσκαλεί τα κράτη-μέλη αλλά αυτό είναι ένα διπλωματικό τρόπο να, να πει κανεί ότι κάνετε ό,τι θέλετε, εμεί δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα να σα εμποδίσουμε ο Μάρκο Φρόντε. Σας ευχαριστώ. Αυτό το πρόγραμμα δράσης μας ικανοποιεί. Σύμφωνα με τους τρεις άξονες, την πρόληψη που είναι πολύ σημαντική, καλύτερη υλοποίηση και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων ε, και ακριβώς θα αναβαθμιστεί αυτό το πρόγραμμα δράσης για να αποκτήσει αποτελεσματικότητα, να αποδώσει αποτελέσματα, δηλαδή και με έναν μηχανισμό παρακολούθησης της πρόοδου αυτού του προγράμματος και να υπάρχουν ε, συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα προς τούτο. Και ε, όλα αυτά δεν ισχύουν σήμερα στο σημερινό πρόγραμμα δράσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά και πρώτα-πρώτα θα πρέπει να δούμε για το Συμβούλιο. Υπάρχει εδώ ένα χάσμα μεταξύ στόχων και προσπαθειών. Ε, τι κάνει η Ευρώπη για το θεματολόγιο. Τι θέλει να πετύχει και τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Εναρμόνιση, συντονισμός, ε, ομοιομορφία στη δράση. Τι γίνεται με το θεματολόγιο και είναι σημαντικό να υπάρχουν κάποιες δομές που να χαρακτηρίζονται ακριβώς από ομοιογένεια, κάτι το οποίο πρόσφατα δεν ισχύει. Α, και στην Ιταλία υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες, κάποια γραφεία τσίτες, αλλά αυτές οι υπηρεσίες κλείσανε γιατί διαλύθηκε η αγροφυλακή, η δασοφυλακή και έτσι οι αρμοδιότητες περάσανε τώρα ε, σε διάφορες άλλες διοκτικές αρχές. Άρα τώρα ο έλεγχος έχει ε, υποβαθμιστεί όσον αφορά αυτό το παρανομό εμπόριο. Τι γίνεται με τις κυρώσεις. Θα πρέπει οι κυρώσεις να γίνουν πιο αυστηρές, να συντονιστούν καλύτερα οι διοκτικές αρχές ούτως ώστε η υποπτία να είναι καλύτερη και επομένως να δρουν αποτριπτικά αυτές οι πιο αυστηρές κυρώσεις κατά του φαινομένου που θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Οπότε χρειάζεται να υπάρξει δέσμευση, στράτευση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Να υπάρξει χρηματοδότηση, να υπάρξει προοικοδότηση. Μιλάμε για προστασία της φύσης και της ε, πανίδας της άγρας. Αλλά έχουμε εδώ την άλλη μεριά τώρα κάποια παρανομή δραστηριότητα. Και επομένως θα πρέπει να δοθεί μάχη σε περισσότερα μέτωπα. Το τελευταίο τώρα είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη πέραν των άλλων να προσπαθήσει περισσότερο και προς τα έξω. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ε, των λαθροκυνηγών. Και είπαμε ότι 3% αυτών ε, κάνουν τη ζωή τους ε, και λένε όμως οι ιδιωτικές αρχές ότι δεν είναι εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την δραστηριότητα. Τη λαθροθυρία δηλαδή. Και όπως είπε ένας συνάδελφος, θα πρέπει να στραφούμε και στο πώς θα μειωθεί η ζήτηση στην αγορά. Μην μιλάμε μόνο για καταπολέμηση του εμπορίου η μείωση των προϊόντων λοιπόν από αυτά τα άγρια είδη. Γιατί πάρα πολλοί εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση χωρίς να ξέρουν ότι πρόκειται περί απαγορευμένης δραστηριότητας. Επομένως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Είναι φιλόδοξο αυτό το σχέδιο και ελπίζω να καταφέρουμε κάτι και όλο αυτό το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μίλλερ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω για μένα που έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση με το Συμβούλιο και την Ολλανδική Προεδρία για το σχέδιο δράση γιατί εδώ τίθεται το θέμα τη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. γιατί τα σημεία, κάποια σημεία του σχεδίου δράση εξαρτώνται από την συμμετοχή των κρατών μελών. Είναι πολύ σωστό αυτό λοιπόν και αυτό που είπε ο κύριο Σερβράντι, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι έτοιμα να αναλάβουν όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά την υποστήριξη του σχεδίου δράσης για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Η χρησιμοποίηση λοιπόν αυτών των κονδυλίων και η παροχή ανθρωπίνων πόρων για την ε, ε, λειτουργία του σχεδίου δράσης είναι απαραίτητη. Ε, για την πρόταση τώρα του κυρίου Τέιλορ, νομίζω και εγώ ότι πρέπει να δούμε το ότι τα ζώα τα οποία είναι προστατευόμενα σε τρίτες χώρες να μην έρχονται στην Ευρώπη με παράνομο τρόπο θα πρέπει να εμποδιστεί αυτό το εμπόριο και επομένως θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και για την προστασία ζώων σε, τρίτη, σε τρίτες χώρες και ίσως μπορούμε να προχωρήσουμε με ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές που ανέφερε το Lacey Act των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν ακόμα στο εμπόριο απειλουμένων ειδών στην Ευρώπη που θα πρέπει να απαγορευτεί. Και αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο πραγματικά αυστηρό και αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Ο Μάκ είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν είναι μπόρεσα να μου να στο σύνολο τη συζήτησης αυτής και της ανταλλαγής απόψεων λόγω κόλλημάτων. αλλά θέλω και εγώ να υπογραμμίσω ότι θέλουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης ώστε να αντιμετωπίσουμε το εμπόριο απειλουμένων ειδών. Αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει εκατομμύρια ευρώ στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος και οδηγεί και σε αστάθεια σε πάρα πολλές ε, χώρες. Υπάρχουν ακόμα και γεωπολιτικά πράγματα, τα γεωπολιτικές πτυχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Θέλω να σας παραπέμψω και στο σχέδιο δράσης για τη βιοπικιλότητα. Υπήρξε η διαμαρτυρία για το γεγονός ότι δεν υπήρξε ένα σύνολο κανόνων για το εμπόριο των ειδών αυτών και θεωρήθηκε αυτό ότι ήταν ένα κενό μέσα στο σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε στο τέλος του Φεβρουαρίου ήταν κάτι το οποίο θεωρήθηκε καλό δεκτό. Πάντα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα βέβαια. Και το θέμα είναι πώς θα μεταφέρουμε την θέλησή μας στην πράξη. Εγώ θα ήθελα να ξέρω από, τον, από την Ολλανδική Προεδρία πώς αντιμετωπίστηκε από τα κράτη-μέλη αυτό το πρόγραμμα και πώς αξιολογείται την πολιτική θέληση των κρατών μελών να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο και να δώσουν ανθρώπινους πόρους και χρήματα για αυτό. Και επίσης σε μια πρόσφατη συνάντηση που οργανώθηκε από τον εισηγητή μας. Υπήρξε μια αναφορά στο νόμο Lacey, το Lacey Act των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανατρέχει στο 1900 και απαγορεύει την εισαγωγή ειδών που προστατεύονται στη χώρα προέλευσής τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπω στο σχέδιο δράσης να υπάρχει. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν αυτό και είναι κάτι το οποίο το συζητά το Συμβούλιο τώρα ή όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θέλει να σχολιάσει. Εάν ναι, τώρα είναι η ώρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη Δευτέρα Ακούσαμε ότι υπάρχει θετική ε, ανταπόκριση από τους βουλευτές και αυτό μας ικανοποιεί. Πρέπει να πω ότι μεγάλο μέρος ε, της εφαρμογής εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη, έχουμε διαβουλεύσει συνεννόηση μαζί τους. Υπάρχει μια επιτροπή με ανταλλαγή ε, πρακτικών, διδασκόμαστε ένας από τον άλλο. Και όσο προχωρούμε και σε ό,τι αφορά την παρουσίαση που έκανα νωρίτερα, ε, δηλαδή για την Νότια Αφρική κτλ. Αλλά και στο άλλο μέτωπο εργαζόμαστε από κοινού με τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τον νόμο λέει, εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι η διάσκεψη σάιτε είναι ε, η νομική πράξη που πρέπει να είναι προτεραιότητα. Εργαζόμαστε με χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν νέες προτάσεις συνεχώς. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο όμως τα κράτη-μέλη έχουν να μας δώσουν παραδείγματα για το ότι υπάρχουν απειλούμενα είδη με μονομένες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από τις σάιτες. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν έχουμε όμως πληροφορίες σε σχέση με τεράστια κενά ενδεχόμενα στην διάσκεψη ΣΑΙΤΕΣ. Ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες ε, μας κάνουν προτάσεις για προσθήκη ειδών ε, στις ΣΑΙΤΕΣ, στα παραρτήματα δηλαδή, και πολλές από αυτές τις προτάσεις στηρίζουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ. Εσείς τώρα από την Ολλανδική Πρόεδρε για να καταλήξετε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ενθαρρυντικό αυτό που πρόκειται από τη συζήτηση σήμερα, ότι δηλαδή και τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι είναι επίγον να αντιμετωπίσει το σημαντικό αυτό ζήτημα. Συμφωνώ ότι έχει γίνει καλή πρόοδος και περιμένω ότι και τη Δευτέρα θα καταστεί σαφέ ότι και το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι καλό βήμα προ τα εμπρό το σχέδιο δράση τη Κομισιόν για την επίλυση αυτών των προβλημάτων που συζητούμε σήμερα. Θα ήθελα τώρα να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα. Βέβαια, πρέπει να καταστήσω σαφέ ότι και εγώ από τη δική μου ιδιότητα έχω κάποια όρια. Δεν μπορώ να ε, ξεπεράσω το ρόλο μου και δεν μπορώ να σχολιάσω πράγματα τα οποία δεν εντάσσονται στο σχέδιο δράση έτσι, πρώτα απ' όλα, ούτε και να μπω σε λεπτομέρειε ε, σε ό,τι αφορά τι 32 δράσει του σχεδίου. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι αυτό που είπα και πριν στην εισαγωγή μου, ότι δηλαδή τη Δευτέρα περιμένω το Συμβούλιο να εκφράσει την υποστήριξή του προ το σχέδιο δράση και τι προτεραιότητε του. Το ίδιο θα κάνει ε, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, αφού είναι ένα και αδιαρρεύτο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει διαφορά επειδή το εγκρίνει το Συμβούλιο περιβάλλοντο. Επίση, συμφωνώ με τι δηλώσει των βουλευτών ότι πολλά εξαρτώνται και από την εφαρμογή αυτών των δράσεων και από πλευρά Συμβουλίου επίση προσβλέπουμε στην εφαρμογή των δράσεων του σχεδίου τη Κομισιόν. Θεωρούμε και εμεί ότι είναι σημαντική η παρακολούθηση, ο έλεγχο τη εφαρμογή των δράσεων. Και η Κομισιόν θα πρέπει να μα τηρεί ενημέρωση για την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή των δράσεων. Κάτι θα λέει και το κείμενό μας της Δευτέρες από αυτού. Δύο λόγια τώρα για ένα θέμα που κάποιος ανέφερε για τις σάιτες, ε, τη 17η διάσκεψη. Είμαστε εν μέσω της προετοιμασίας για αυτή τη διάσκεψη. Θα είναι η πρώτη διάσκεψη στην οποία συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέες προκλήσεις λοιπόν και νέες ευκαιρίες. Συνεργαζόμαστε στενά με τη Σλοβακική Προεδρία, την επόμενη δηλαδή από εμάς και την Κομισιόν, για να παρουσιάσουμε μια κοινή θέση στην διάσκεψη της ΆΙΤΕΣ και ελπίζουμε να μας στηρίξει και το δικό σας ε, ψήφισμα, που τώρα μόλις το διάβασα και σίγουρα θα μας υποστηρίξετε ε, σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και οποίες θα περιλαμβάνουν λιοντάρια, καρχαρίες, ελέφαντες και πάγκαλινς να ε, προστατεύονται. Είναι ζώα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι σύμβολα. Υπάρχουν και άλλα όπως η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς και της τροπιοθυρίας σημαντικά και αυτά. Πρώτο βήμα λοιπόν για την υλοποίηση του σχέδιου δράση κατά πολέμηση του λαθρεμπορίου άγριων ειδών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπόλ, φαντάζομαι και αυτό θα το πούμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη Δευτέρα, κατάσταση νομίζω είναι σαφή. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, εκφράσουν τις προτεραιότητές τους στην Europol, να τις δώσουν δηλαδή πληροφορίες και να τις πούν ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας. Είναι απαραίτητο για να δώσει την απαραίτητη συνέχεια η Europol, γιατί βασίζει την δράση της στις πληροφορίες και στις προτεραιότητες που παίρνει από τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ζητήσουμε και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αν πια είναι όλα τόσο σημαντικά, θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό και η Ευρωπόλ. Νομίζω απάντησα στα περισσότερα ερωτήματα που σημείωσα τουλάχιστον και που μπορούσα να απαντήσω άμεσα. Εν κατακλείδη, να πω ότι προσβλέπουμε στη συνεδρία της Δευτέρας, που ελπίζουμε εκεί το Συμβούλιο Περιβάλλοντος να δείξει πόσο δεσμευμένο είναι στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και περιμένουμε να έχουμε βέβαια και περαιτέρω συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή σας όλους ιδιαίτερος και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που μου δώσετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για τις απαντήσεις και τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Ε, υπάρχει κάτι τα διάφορα. Άρα το επόμενο σημείο είναι η δεξαμενή επόμενη συνεδρία που θα γίνει την 21η Ιουνίου στι Βρυξέλλε. Καλή σα ημέρα, γεια σας.